La seduta è ripresa. Επαναλαμβάνεται η σύνοδος. Να σας ενημερώσω για τα αποτελέσματα της δεύτερης ψηφοφορίας. Εψήφισαν 704. Λευκά ή άκυρα 37. Έγκυρες ψήφοι 667. Απόλυτη πλειοψηφία, απαραίτητη, 334 ψήφοι. Οι υποψήφοι έλαβαν τις εξής ψήφους. Κέλλερ, 119. Ρέγκο, 43 ψήφοι. όλοι. 345. Ζάχραντιλ. 160. Ο κύριος Σασόλη έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία των ε, ε, έγκυρων ψήφων. Ο κύριο Σασόλη είναι ο νέο πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου. Τον συγχαίρω για την εκλογή του. Με κάθε ε, ευχή για επιτυχία στην θητεία του. Παρακαλώ, μπορείτε να αναλάβετε την Προεδρία του Ευρωκοινοβουλίου. συνάδελφοι, φίλοι μου, εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων, των κυβερνήσεων, γυναίκες και άνδρες της διοίκησης του Κοινοβουλίου. Θα καταλάβετε όλες και όλοι τη συγκίνησή μου αυτή τη στιγμή, τη στιγμή που αναλαμβάνω την Προεδρία του Ευρωκοινοβουλίου. Με επιλέξατε εσείς για να εκπροσωπώ τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα το όργανο αυτό που έχει άμεσου δεσμούς με τους πολίτες και καθήκον του είναι να του προασπίζεται και να τους εκπροσωπεί. Να θυμόμαστε πάντοτε ότι η ελευθερία μας είναι καρπός της δικαιοσύνης που καταφέραμε να αποκτήσουμε και της αλληλεγγύης που μπορούμε να προωθούμε. Να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Αντώνιο Ταγιάννη για το έργο του σήμερα, για τη μεγάλη του αφοσίωση και την πίστη που έδειξε στον, ε, ε, στο Ευρωκοινοβούλιο ως θεσμικό όργανο. Να καλωσορίσω τους βουλευτές που έλαβαν τη διαπίστευσή τους, ε, γυναίκες και άντρες, τις γυναίκες κυρίως που είναι το 40% του συνόλου ε, των βουλευτών στην Ευρωβουλή. Είναι πολύ καλό το αποτέλεσμα, αλλά θέλουμε περισσότερες. σε αυτή τη φάση, μετά από μια έντονη προεκλογική εκστρατεία και στην έναρξη μιας νέας κοινοβουλευτικής θητείας, Έχουμε να αναλάβουμε μεγάλες ευθύνες. Κανείς δεν μπορεί να αρκεστεί στο να παραμένουμε σε όσα έχουμε κεκτημένα. Έχουμε το εκλογικό αποτέλεσμα, το βλέπουμε με τη σύνθεση αυτής της Ευρωβουλής, αλλά ζούμε ε, καμπές ε, τεράστιες ε, στον κόσμο μας. Η ανεργία των νέων, οι κλιματικές αλλαγές, η τεχνολογική επανάσταση, η νέα ψηφιακή ε, εξέλιξη είναι τεράστιες προκλήσεις που για να τις διαχειριστούμε θα πρέπει να το κάνουμε με καινούριε ιδέες, με, με την τόλμη να συνδυάσουμε μεγάλη, την μεγάλη σοφία και την ε, τόλμη που θα πρέπει να δείξουμε. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε το πνεύμα των ιδρυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτών που ε, μπόρεσαν τότε να αφήσουν πίσω τους τις εχθροπραξίες και το κλίμα του πολέμου, ε, μην ξεχνώντας τις καταστροφές του εθνικισμού. Ε, έτσι δημιουργήθηκε αυτό το εγχείρημα για να συνδυάσουμε την ειρήνη, τη δημοκρατία, τα δικαιώματα, την ανάπτυξη και την ισότητα. Αυτούς τους μήνες είδαμε ότι το εγχείρημα της Ευρώπης υποβαθμίστηκε αρκετά. Υπήρξαν διαφορετικές απόψεις και συγκρούσεις. Αυτές ε, είναι οι θλιβερότερες αναμνήσεις της ιστορίας μας. Οι πολίτες έδειξαν όμως ότι πιστεύουν, πιστεύουν ακόμα σε αυτήν την ε, εξαιρετική ε, ιδέα και αυτό το εγχείρημα. Ότι μπορούμε να βρούμε απαντήσει στι διεθνεί προκλήσει, ε, αυτέ που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να βρούμε τη δύναμη να ξεκινήσει ξανά η διαδικασία ολοκλήρωση, να αλλάξουμε την ενωσή μα και να γίνει ικανή να ανταποκριθεί με τρόπο ακόμα πιο αποφασιστικό στις απαιτήσεις των πολίτων, να δώσει, πολίτων, να δώσει πραγματικές απαντήσεις στις ανησυχίες τους, την ε, ε, δική τους αίσθηση δυσφορίας ότι τα πράγματα κάπως έχουν ξεφύγει από τη σωστή πορεία. Πρέπει να θυμηθούμε τις ιδρυτικέ αξίες της ελευθερίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης. Αυτά πρέπει να τα εκφράζουμε καθημερινά, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, θα πρέπει πιο συχνά να σκεφτόμαστε σε τι κόσμο καλούμαστε να ζήσουμε και τι ελευθερίες ε, είμαστε σε θέση να απολαμβάνουμε. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε εμείς πρώτοι, γιατί άλλοι ανατολικά μας, δυτικά μας, νότια, ε, δεν καταλαβαίνουν, δεν θέλουν να παραδεχτούν ότι αυτό που μας διακρίνει μας κάνει απλώς διαφορετικούς, όχι καλύτερους, διαφορετικούς. Ως Ευρωπαίοι είμαστε υπερήφανοι για την διαφορετικότητά μας και το επαναλαμβάνουμε. Στην Ευρώπη καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να καταστρέφει τις ιδρυτικές αξίες της Ευρώπης. Την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Οι αξίες μας αυτές μπορούν και να δείξουν και το κατά πόσο να αξίζουν τον κόπο οι πολιτικές μας στην Ευρώπη. Κανείς δεν μπορεί να φημώνει τους ε, ε, αντιπάλους του οι κυβερνήσεις που εκπροσωπούν ε, το λαό, που κυβερνούν τους λαούς της Ευρώπης, είναι αποτέλεσμα ελεύθερων εκλογών, νόμιμων εκλογών. Κανείς δεν μπορεί να καταδικάζεται για, την για το θρησκευτικό του δόγμα, για τις φιλοσοφικές του απόψεις, για την ιδεολογία του. Ε, θα πρέπει τα παιδιά μας να μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα, να ε, σπουδάζουν όπου θέλουν, να αγαπούν χωρίς όρια και σύνορα. Κανείς Ευρωπαίος δεν μπορεί να ταπεινώνεται ή να περιθωριοποιείται για τη σεξουαλικό του προσανατολισμό. Θα πρέπει σε αυτόν τον ευρωπαϊκό χώρο να υπάρχουν διαφορετικά συστήματα ταυτόχρονα, κοινωνικής προστασίας. Αυτό είναι μέρος της ταυτότητάς μας και το οικονομικό και ε, το κοινωνικό μας μοντέλο πρέπει να, ε, να, να ανανεωθεί. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ανάπτυξη, κοινωνικές εξελίξεις και σεβασμό για το περιβάλλον. Όλα αυτά να ε, διευκολυνθούν. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια και να δώσουμε προοπτικές στους νέους μας, να ξεκινήσουμε νέες επενδύσεις, βιώσιμες και να ενισχύσουμε τη διαδικασία σύγκληση μεταξύ των περιφερειών μα και των διαφορετικών περιοχών τη Ευρώπη. Η ψηφιακή επανάσταση αλλάζει τελείω τη φυσιογνωμία μα και τον τρόπο ζωή μα, το πώ παράγουμε και καταναλώνουμε. Χρειαζόμαστε λοιπόν κανόνε, κανόνε που να συναρθρώνουν τι τεχνολογικέ εξελίξει με τι ε, ανάγκε των επιχειρήσεων αλλά και των εργαζομένων και των ανθρώπων. Οι κλιματικέ αλλαγέ μα αφήνει έκθετου σε τεράστιου κινδύνου που πλέον του γνωρίζουμε, ε, χρειάζονται επενδύσει και καθαρέ τεχνολογικέ λύσει για να ανταποκριθούμε στι ε, απαιτήσει των νέων που βγήκαν στου δρόμου. Κάποιοι βρίσκονται και σε αυτή την αίθουσα για να μα θυμίζουν ότι δεν υπάρχει άλλο πλανήτη για να ζήσουμε. Έναν έχουμε θα πρέπει να εργαστούμε για να υπάρχει ισότητα των φύλων, για να αναλαμβάνουν περισσότερε αρμοδιότητε οι γυναίκε στι κορυφαίε θέσει και τα αξιώματα τη πολιτική, τη κοινωνία και τη οικονομία. Κυρίε και κύριοι, αυτό θα είναι το επισκεπτήριό μας για έναν κόσμο που δεν έχει κανόνες, αλλά πρέπει να έχει. Και θέλουμε να βοηθήσουμε να διέπεται η λειτουργία του από κανόνες. Όλα αυτά δεν έχουν συμβεί τυχαία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένα τυχαίο προϊόν της ιστορίας. Εγώ είχα έναν πατέρα που στα 20 του ε, πολέμησε εναντίον και με άλλους Ευρωπαίους. Και είμαι, είχα μια μητέρα που και εκείνη στα 20 της εγκατέλειψε την αιστεία τη και αναγκάστηκε να ζήσει σε διαφορετική οικογένεια. Αυτή είναι η ιστορία και πολλών από τις δικές σας οικογένειες. Και νομίζω ότι αν συνδυάσουμε ο καθένα τη δική του εμπειρία, τη δική του ιστορία και καθίσουμε μπροστά σε ένα ποτήρι εμπειρία να τα διηγηθούμε ένα στον άλλο, θα αντιληφθούμε ότι είμαστε παιδιά και εγγόνια, αλλά ε, όχι ενός τυχαίου περιστατικού της ιστορίας. Η ιστορία μας όμως έχει γραφτεί με πόνο, με το αίμα των νέων Βρετανών που έχασαν τη ζωή τους στην Ορμανδία ή με την επιθυμία ελευθερίας με την ε, ε, με το φόβο και την, τις, τις διαμαρτυρίες για ελευθερία όσων ήταν στις πλατείες της Βαρσοβίας, των ε, όσων ε, καταπιέστηκαν με τα όπλα στις χώρες της Ανατολής. Εδώ χρειάζεται να διεκδικήσουμε την αξιοπρέπεια, την αξιοπρέπεια και να ε, μην εγκαταλείψουμε την ανθρωπιά. Δεν μπορεί η αν υπακόει να θεωρείται αρετή. Δεν είμαστε λοιπόν ατύχημα της ιστορίας. Είμαστε παιδιά και γκόνια όσων κατάφεραν να βρουν μια απάντηση, ένα αντίδοτο σε αυτήν την εθνικιστική ε, υποβάθμιση, ε, αυτό το βρικαλαίο δημιούργημα που προέκυψε στην ιστορία μας. Είμαστε όλοι Ευρωπαίοι και λατρεύουμε τις χώρες μας. Ο εθνικισμός όμως που γίνεται ιδεολογία και ιδεολειψία δημιουργεί θανάσιμους κινδύνους, ιούς που μπορεί να δημιουργήσουν και ε, καταστροφικές ε, εχθροπραξίες και αντιπαραθέσεις. Δεν χρειαζόμαστε διχασμούς, συνάδελφοι. Γι' αυτό χρησιμεύει η πολιτική. Χρειάζονται τα ευρωπαϊκά κόμματα, ευρωπαϊκές ομάδες που θα πρέπει να είναι ανάχωμα για να προασπιστούμε την δημοκρατία μας θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μα. Η θητεία αυτή θα πρέπει να ενισχύσει τι διαδικασίε, να καταστήσει το Ευρωκοινοβούλιο πρωταγωνιστή. Πρωταγωνιστή σε μια ε, αληθινή ευρωπαϊκή δημοκρατία. Δεν ξεκινάμε όμω από το μηδέν. Δεν ξεκινάμε από το τίποτα. Η Ευρώπη βασίζεται στα θεσμικά της όργανα, που παρόλο που είναι ατελή, παρόλο που χρειάζονται μεταρρύθμιση, μας έχουν εγγυηθεί ως τώρα την ελευθερία μας, την ανεξαρτησία μας με τα θεσμικά μας όργανα θα πρέπει να απαντήσουμε και σε όσους έχουν αναλάβει το ρόλο να μας διχάσουν, να μας χωρίσουν. Θα πρέπει λοιπόν στην αίθουσα αυτή, στην αρχή της θητείας να πούμε ότι θα είναι θεματοφύλακα στις ανεξαρτησίες των Ευρωπαίων πολιτών το Κοινοβούλιο. Αυτοί είναι οι μόνοι που έχουν την ευθύνη να καθορίσουν το πεπρωμένο τους. Κανείς δεν μπορεί για λογαριασμό τους. Κανείς, τους, κανείς στη θέση τους ή αντί ημών των ιδίων στην αίθουσα αυτή μαζί με τόσους συναδέλφους, γυναίκες και άντρες, πολύ πυρούς, και καθώς και πολλούς καινούριου βουλευτές, τους οποίους καλωσορίζω θερμά, να πω ότι διάβασα πολλά από τα βιογραφικά τους και είμαι πεπισμένος ότι πρόκειται για παρουσίες θετικότατες. Το 63% αυτού του Ευρωκοινοβουλίου αποτελείται από βουλευτές που εξελέγησαν για πρώτη φορά. Πολλοί από αυτούς είχαν κοινωνικές δραστηριότητε, έχουν πολλά προσόντα, μεγάλη επαγγελματική πείρα. Πολλοί έχουν ασχοληθεί και με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αυτό είναι ένα πεδίο στο οποίο θα πρέπει να κάνει βήματα προόδου η Ευρώπη. Διότι έχουμε νέα φαινόμενα να αντιμετωπίσουμε. Την μετανάστευση, κυρίως. Εδώ θα πρέπει να ε, μην γίνεται πάντοτε αυτή η διελκυστίδα μεταξύ των κυβερνήσεων που κάθε φορά που κάτι συμβαίνει και είμαστε προετοίμαστοι. Το λέω για το Συμβούλιο. Ε, εδώ θα πρέπει να γίνουμε φόρουμ για να συζητηθεί μεταρρύθμιση του κανονισμού του Δουβλίνου. Στην ε, Ολομέλεια έχει προταθεί αυτό ήδη από την προηγούμενη θητεία με τεράστια πλειοψηφία. Θα πρέπει λοιπόν ως χρέος να το πράξουμε αυτό για τους Ευρωπαίους πολίτες. Ζητούν οι πολίτες μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Αλλά το οφείλουμε και σε αυτούς τους ε, ε, καημένους ανθρώπους που δεν θέλουμε να χάσουν την αίσθηση ανθρωπιάς ε, που πρέπει να επιδείξουμε. Κύριοι του Συμβουλίου, είναι η απόφαση στα χέρια σας δεν μπορείτε να απεκδίεστε των ευθυνών σα. Ούτε μπορείτε να βάλετε τι αποφα... τις αποφάσεις τη δυσπιστία απέναντι στην ενωσή μα. Οι πολίτε αναρωτιούνται με, με κάθε κατεπήγον που συμβαίνει πού είναι η Ευρώπη, τι κάνει αυτή η Ευρώπη. Αυτό θα είναι ακριβώ και το μεγαλύτερο τεστ, η μεγαλύτερη δοκιμή για μα, για να αντιμετωπίσουμε τι δυσπιστίε και τι ε, εθνικέ εγωπάθειε. Θα πρέπει λοιπόν το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή να αναλάβουν αυτό το καθήκον, να αποκριθούν με μεγαλύτερη τόλμη στις απαιτήσει των νέων μας, που ζητούν με ηχηρέ φωνέ να ξυπνήσουμε, να ανοίξουμε τα μάτια, να σώσουμε ανθρώπινε ζωές. Απευθύνομαι λοιπόν σε εκείνου. Να θεωρείτε αυτό το κοινοβούλιο που σήμερα ξεκινά τη νέα του θητεία ω το δικό σα σημείο αναφορά. Βοηθάτε μας Βοηθάτε μας να είμαστε και πιο τολμηροί για να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει τη αλλαγή που έχουμε μπροστά μα. Διαβεβαιώ Διαβεβαιώ το Συμβούλιο και τι εναλλασσόμενε προεδρίε ότι θα πρέπει να υπολογίζουν στην ε, υποστήριξή μα και τη συνεργασία μα. Το ίδιο και στην Επιτροπή με τον νέο τη Πρόεδρο. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να ανασχεδιάσουν του εαυτού του. Δεν θα υπάρξουμε πρόσκομα στην ε, οικοδόμηση μιας ε, πιο ενωμένης Ευρώπης. Και προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θέλω να απευθύνω και χαιρετισμό εκ μέρου του ε, μέσω εκείνου στου αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων. Ε, στους 28 που αποτελούν τη Μεγάλη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι 28 κράτη. Μικρά ή μεγάλα είναι το καθένα ένας θησαυρό μοναδικός στον κόσμο. Όλοι έχουν μακρά ιστορία. Όλοι έχουν πολιτισμό, γλώσσα, τέχνη, φύση, τοπία, ποίηση. Αυτά δεν μπορεί να τα μιμηθεί ούτε να τα παραχαράξει κανείς. Είναι ε, περιουσιακά στοιχεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς που όλοι σεβόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν όταν θα σας επισκεφθώ εξ ονόματος των βουλευτών ουδέποτε θα ξεχάσω ότι μπροστά στις σημαίες και τους εθνικούς ύμνους θα πρέπει να αποτίσουμε φοροτιμής σε όσους δείχνουν τον απαραίτητο σεβασμό εδώ σε αυτή την αίθουσα. Το αντίθετο για όσους δεν τον δείχνουν. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να χαιρετήσω και τους Βρετανούς βουλευτές και θα τους έλεγα να σκεφτούν καλά το Brexit, το Βερολίνο, ε, το Παρίσι, τη Ρώμη, τη Μαδρίτη. Δεν μπορούμε να τα σκεφτούμε μακριά από το Λονδίνο. Μας πονάει αυτό. Σκεφτείτε το. Με κάθε σεβασμό που οφείλουμε βεβαίω στην επιλογή των Βρετανών πολιτών. Για μας τους Ευρωπαίους είναι ένα πολιτικό βήμα που θα πρέπει να γίνει με ορθολογισμό, διάλογο και σε πνεύμα φιλικό. Και πάντοτε με πλήρη σεβασμό των κανόνων και των αντιστοίχων δικαιωμάτων πρωτοβουλία που έχουν η ΜΕΝ και η ΔΕ. Χαιρετίζω και του εκπροσώπου των κρατών που θέλησαν και έχουν υποβάλει τι προσχώρησει προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την εξέταση αυτή τη ε, επιλογή. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ βολικό να είναι κανεί μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι διαδικασίε προσχώρηση έχουν κινηθεί και το Κοινοβούλιο πολλέ φορέ έχει δηλώσει την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί ω τώρα. Καλή τύχη λοιπόν και σε όλη τη δίκηση του συνεργάτε αυτού του Κοινοβουλίου. Έχουμε θέσει ένα στόχο από την προηγούμενη θητεία. Να γίνει το Ευρωκοινοβούλιο ο οίκος της δημοκρατίας για την Ευρώπη. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μεταρρύθμιση, ε, διαφάνεια, καινοτομία. Πολλά αποτελέσματα τα έχουμε πετύχει ήδη και για τον προπολογισμό. Αλλά σε αυτήν την θητεία θα πρέπει να έχουμε μια εντονότερη όθηση. Και για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε περισσότερο διάλογο μεταξύ βουλευτών και διοίκηση. Δική μου ευθύνη θα είναι να το διασφαλίσω και αυτό. Συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, η Ευρώπη έχει ακόμα πολλά να πει, αρκεί να τα πούμε μαζί. Εσείς όλοι ε, και εμείς όλοι μαζί. Θα πρέπει η πολιτική να τεθεί στην υπηρεσία των πολιτών μας και να πολεμήσουμε, να ακούσουμε τις επιθυμίες, τους φόβους τους και την οργή τους, αλλά πάνω από όλα τις ανάγκες τους. Είμαι βέβαιος ότι όλοι σας θα μπορέσετε να συνεισφέρετε τα μέγιστα σε μια καλύτερη Ευρώπη η οποία θα δημιουργηθεί με εσά, με εμά, αρκεί να εργαστούμε με την καρδιά μας και με όλη μας την ε, φιλοδοξία. Grazie, allora cominciamo subito a lavorare. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε αμέσω στη δουλειά. Εάν οι πρόεδροι των ομάδων θέλουν κάτι να πούν, να εκφραστούν, τώρα είναι η στιγμή να το κάνουν. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα στο όνομα των της ε, πολιτικής μου ομάδας να σας συγχαρώ. Ε, περιμένουμε να δούμε να πραγματοποιείτε αυτά που μόλις είπατε. 201 ε, εκατομμύρια άτομα συμμετείχαν στις ευρωεκλογές και έτσι έχουμε λάβει εμείς οι βουλευτές την εντολή μας. Έχετε αναλάβει μεγάλη ευθύνη και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα σας ε, εύχεται καλή επιτυχία το, ε, τα επόμενα δυόμιση χρόνια. Ε, μας έχετε στο πλευρό σας τις προσπάθειές σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Ιράτσα Γκαρσία Πέρες. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκ μέρους της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θα ήθελα να ξεκινήσω με συγχαρητήρια προς τον πρόεδρο σας όλοι για τις νέες ευθύνες που αναλαμβάνει. Τίποτα δεν μπορεί ε, να περιπίσει περισσότερη τιμή και περηφάνεια σε έναν Ευρωβουλευτή από τη θέση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του θεσμικού οργάνου που εκπροσωπεί την ε, κυριαρχία των πολιτών. Εκπροσωπούμε εδώ άνδρες και γυναίκες που θέλουν να οικοδομήσουν μια περισσότερη, ισχυρότερη και καλύτερη Ευρώπη. Αναπόκειται σε εμά λοιπόν να δώσουμε την απάντηση που περιμένουν από εμά οι πολίτε. Να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη του στο ευρωπαϊκό σχέδιο. Έχουμε μία πενταετία ενώπιον μα για να συνεργαστούμε ε, μεταξύ μας με του Ευρωβουλευτέ, άνδρε και γυναίκε, και για να ενισχύσουμε αυτό το σχέδιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, για να κάνουμε μια Ευρώπη των πολιτών, μια Ευρώπη των δικαιωμάτων και των αρχών, μια Ευρώπη τη ισότητα και τη δικαιοσύνη. Και να πόκεται στα χέρια μα να το καταφέρουμε. Ε, μπορείτε να βασιστείτε στην αμέριστη υποστήριξη και συνεργασία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Γιατί η δική του μοίρα θα είναι η μοίρα και η τύχη το πεπρωμένο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το πεπρωμένο των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ κύριε Πέρες. Ο πρόεδρος Τσόλος έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας συγχαρώ για την εκλογή σας σήμερα. Και είμαι βέβαιος ότι όπως έδειξαν και χθεσινές συζητήσεις θα συνεχίσουμε την πολύ καλή συνεργασία που ξεκινήσαμε. Και μάλιστα ε, οι φετινές ευρωεκλογέ έδειξαν ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες εξακολουθούν να έχουν μεγάλες προσδοκίες από το ευρωπαϊκό σχέδιο και γι' αυτό η τρέχουσα κοινοβουλευτική θητεία θα πρέπει να ανανεώσει αυτό το σχέδιο. Και οι διαβουλεύσεις στο Συμβούλιο έχουν δείξει ότι χρειάζεται πραγματισ... πραγματισμός, ρεαλισμός για αυτή την ανανέωση, την αναζωογόνηση. Και αυτή η αναζωογόνηση δεν θα προέλθει ούτε από το Συμβούλιο ούτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από εμά θα πρέπει να εκπορευτεί, γιατί εμεί είμαστε η φωνή των Ευρωπαίων πολιτών. Εμεί ενσαρκώνουμε αυτή την αναζωογόνηση που χρειάζεται το ευρωπαϊκό σχέδιο. Και σα διαβεβαιώ ότι η ομάδα μα, το Renew Europe, η ανανέωση τη Ευρώπη, θα είναι ένα πολύ καλό εταίρο. Και θα ήθελα να οργανώσουμε μαζί με όλου του Ευρωπαίου εταίρου μια συνδιάσκεψη για το μέλλον τη Ευρώπη για να δούμε πώς θα φέρουμε τους πολίτες μας, τους συμπολίτες μας πιο κοντά στο ευρωπαϊκό σχέδιο. Γιατί δεν πρόκειται οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις να αποφασίσουν ποιος θα βρεθεί επικεφαλής σε ηθήνουσες θέσεις στην Ευρώπη. Οι πολίτες θα πρέπει να δίνουν τη γνώμη τους και εμείς στηρίζουμε ένα τέτοιο διάβημα. Αυτό θα κάνουμε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε. Μαζί, όλοι μαζί, από κοινού, γιατί θα πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βελτιώσει τη σχέση των Ευρωπαίων πολιτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σόλος. Κυρία Κέλλερ. Um, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Συγχαρητήρια. Ε, προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί σας. Ε, τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου είναι ακριβώς αυτό που θα πρέπει να συζητήσουμε εδώ, διότι μέχρι τώρα ως Κοινοβούλιο πάντα προωθούσαμε τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου, διότι αυτό σημαίνει αύξηση των δικαιωμάτων και των πολιτών. Αλλά τώρα ε, αμφισβητείται αυτή η θέση. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να μην εγκαταλείψουμε τον αγώνα, να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να βελτιώσουμε και να αυξήσουμε την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Αυτό είναι το έργο μας και, και δεν επιτρέπεται να εγκαταλείψουμε τον αγώνα αυτό θα πρέπει να στηρίξουμε την ιδέα ότι ε, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα έπρεπε να είναι κάποιος από ε, τους κορυφαίους υποψήφιους, τους Spitzkandidaten. Επίσης θέλουμε ε, υπερεθνικά ψηφοδέλτια. Θα πρέπει επίσης να εργαστούμε πάνω στο θέμα της διαφάνειας εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Θυμάστε τα ψηφίσματα που είχαμε ε, κατά την προηγούμενη θητεία σχετικά με την επανεμπόδιση και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης που δυστυχώς είναι πρόβλημα και εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα σας παρακαλούσα, σας καλώ να ε, ε λάβετε σοβαρά υπόψη σας σε αυτά τα ψηφίσματα, διότι ε, πρέπει να σταθούμε στο πλευρό των θυμάτων. Επίσης, κύριε Πρόεδρε, ένα μέλος των Πρασίνων σήμερα δεν ε, ήταν σε θέση να ε, παρευρεθεί ε, διότι δεν έχει υποβάλει το όνομά του το κράτος μέλος παρότι εξελέγει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βρίσκεται είναι απόν σήμερα χωρίς να φταίει ο ίδιος. Σας παρακαλώ λοιπόν να λάβετε υπόψη σας τα δικαιώματα του κυρίου Κέρας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριος Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχετε πλέον το καθήκον και το φορτίο να καθοδηγείτε αυτήν την Ολομέλεια και το Κοινοβούλιο, το θεσμικό μα όργανο, από τη δύσκολη στιγμή. Τη στιγμή που η απόσταση μεταξύ Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και Πολιτών είναι στην, ε, στο ύψιστο σημείο. Ε, δεν έχουμε καταφέρει να δώσουμε στου πολίτε να καταλάβουν ότι είναι κοντά του τα θεσμικά όργανα τη Ευρώπη. Εκτιμώ τα λόγια που χρησιμοποίησατε και στην αρχική σα ομιλία και στην παρουσίασή σα προηγουμένω. και μερικέ από τις έννοιε που αναπτύξατε τι συμμερίζομαι πλήρως. Είπατε ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να γίνει αυτό ο οίκο οίκο δημοκρατίας για την Ευρώπη. Μιλήσατε για δικαιώματα, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, μιλήσατε για το σεβασμό, για τις διαφορετικές ιδέες δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε στην ομάδα μας, την ομάδα της ταυτότητας και της δημοκρατίας. Όμως κάποια από αυτά αντιφάσκουν με όσα είχατε πει πριν από μερικές μέρες για την ανάγκη να υπάρξει ε, κάποιο είδους περιοριστικό μέτρο, ε, κάποιο είδους ε, κορδόν σανιτέρ, όπως λέμε σε άλλες γλώσσες, για όσους εδώ αμφισβητούν την ε, αξία της δημοκρατικής εκπροσώπησης σε αυτό το κοινοβούλιο και θα πρέπει να δούμε ξανά την πρόσβασή του στο κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι θα πρέπει αυτά που είχατε πει στην ομιλία σας και τα οποία συμμεριζόμαστε να ακολουθούνται τις ανάλογες πράξεις. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να γίνει και σε αυτήν την αίθουσα, αν θέλετε αυτός ο οίκος να γίνει οίκος της δημοκρατίας, αν θέλετε πραγματικά να σεβαστείτε τη βούληση των Ευρωπαίων πολιτών που έδωσαν ε, σε αυτό το κόμμα και την ομάδα μας ε, εκατομμύρια ψήφου, θα πρέπει να έχετε μια επικοδομητική προσέγγιση και να στηρίξετε του υποψηφίου μα για τι διάφορε αρμοδιότητε που θέλουμε να αναλάβουν. Γιατί και οι πολίτε έχουν δικαίωμα να εκπροσωπηθούν και τα δικά του ιδεώδη να εκφράζονται και σε αυτό το κοινοβούλιο. Σα εύχομαι καλή τύχη και ελπίζω πραγματικά τα λόγια σα να ακολουθούνται από τι ανάλογε πράξει. Αλλιώ δεν μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατικό θεσμικό όργανο. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα θεσμικό όργανο που σέβεται τι διαφορετικέ απόψει και τι άλλε ιδεολογίε. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα όργανο που ε, ε, ακολουθεί την επιθυμία των πολιτών για αλλαγή. Ευχαριστούμε κύριε Τζάνι. Ο κύριος Λεντούπτκο. Ο κύριος Φίτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εγώ θέλω να ενώσω τη φωνή μου εκ των συντηρικών και μεταρρυθμιστών ε, στι φωνέ όσων εξέφρασαν ευχές για τη δουλειά σας. Η δική μου αξιολόγηση είναι σαφώς θετική για όσα έχετε κάνει Παρά βεβαίω την πολιτική απόσταση που ε, μας χώρισε και φάνηκε και από την ψηφοφορία. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Ως ομάδα έχουμε διαφορετική τοποθέτηση για πολλά από τα ζητήματα που έχουν τεθεί και θα τεθούν προς συζήτηση στην αίθουσα αυτή και ε, θέλουμε η Ολομέλεια να επιστρέψει στην, στο πρωταγωνιστικό ρόλο που θα πρέπει να έχει για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων που ανήκονται μπροστά μα. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε διαφορετική μέθοδο. Όχι συμφωνίε που ε, γίνονται και κλεισμένα των θυρών και μετά έρχονται και ανακοινώνονται εδώ σε μια αίθουσα ολομέλεια. Θα πρέπει τα πράγματα να αλλάξουν. Να αλλάξει το κοινοβούλιο και στον τρόπο τη διοργανωσή του και στι επιλογέ του και να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στο ρόλο των κρατών μελών. Να αναλάβουν δράση για τα μεγάλα ζητήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Δεν θα σα λείψει λοιπόν η δική μα συνεισφορά οπωσδήποτε, αλλά η συνεισφορά μα θα είναι προσπάθεια ε, νέα εξισορρόπηση τη ε, προσέγγιση μας. Πρέπει να ε, αναλάβουμε τις νέε αρμοδιότητες που καλούμαστε να αναπτύξουμε στο νέο ιστό της Ευρώπης. Ευχαριστούμε κύριε Φίτο. Ο κύριος Σίρντεβαν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια και από μένα για την εκλογή σας. Στην ε, ομιλία σας αναφερθήκατε σε σημαντικά πολιτικά εγχειρήματα, ε, μερικά από τα οποία συμμεριζόμαστε και εμείς ε, ως αριστερή ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Χρειαζόμαστε όμως μια κοινή δημοκρατική βάση. Ένα αίτημα, ένα αίτημα προς εσάς να συνεργαζόμαστε με πιο διαφανή τρόπο μεταξύ μας και να λαμβάνονται υπόψη και τα δικαιώματα των μικρότερων πολιτικών ομάδων του Κοινοβουλίου. Ε, προσβλέπουμε στην συνεργασία πάνω σε προοδευτικά έργα και ελπίζουμε να έχουμε και μια προοδευτική ανταλλαγή απόψεων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους Προέδρους των πολιτικών ομάδων για τις παρεμβάσεις τους και τώρα προχωρούμε στην συγκρότηση σώμα των πολιτικών ομάδων. Κάτι που πρέπει να γίνει στην αρχή της κοινοβουλευτικής θητείας. Αυτή είναι η εξή ανακοίνωση. Δημιουργήθηκαν οι εξή πολιτικές ομάδες. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, 182 βουλευτές η Προοδευτική Συμμαχία Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωκοινοβούλιο, 154 βουλευτές, η ομάδα Renew Europe, 108 βουλευτές, Πράσινη Ελεύθερη Συμμαχία για την Ευρώπη, 74 βουλευτές. Ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία, 73 βουλευτές. Ομάδα Συντηρητικών και Μεθαρρυθμιστών της Ευρώπης, 62 ε, βουλευτές. Συνόσπονδη Ομάδα της ε, Ενωμένης ε, Ευρωπαϊκής Αριστεράς και Βόρειας Αριστεράς, 41 βουλευτές και 57 μη εγγεγραμμένοι βουλευτές. Οι δηλώσει για τη συγκρότηση σε σώμα των ε, πολιτικών ομάδων βάσω του άρθρου 33, εδάφιο 5 του εσωτερικού κανονισμού θα προσαρτηθούν στα πρακτικά αυτή τη συνόδου. Περνούμε τώρα στην ημερήσια διάταξη, το τελικό σχέδιο ημερήσια διάταξη όπω έχει κρυφθεί από τη διάσκεψη των Προέδρων στι 30 Ιουνίου βάσει του άρθρου 127 έχει διανεμηθεί. Ανακοινώνω ότι δεν έχω λάβει καμία αίτηση για αλλαγή στην, στο τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης, οπότε θεωρούμε ότι εγκρίνεται. Περνάμε σε μια πρώτη ψηφοφορία. Την αριθμητική σύνθεση των μόνιμων επιτροπών γνωρίζετε την πρόταση. Υπέρ, διανάταση ισχυρό, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε στην εκλογή των αντιπροέδρων. Εκλογή των αντιπροέδρων του Κοινοβουλίου. Για την εκλογή των αντιπροέδρων, προθεσμία για την υποβολή υποψηφιωτήτων μέχρι τις 14 και 45 σήμερα. Η ψηφοφορία θα γίνει στις 15 και 45. Οι υποψηφιότητες έχουν αποσταλεί στους υπεύθυνους του γραφείου 121 Open Space της Προεδρίας ε, στο Louis Φάις. Η σύνοδος διακόπτεται. Θα συνεχίσουμε στις 3. Ευχαριστώ. 15 και 45 για την ακρίβεια. Ευχαριστώ. Ναι. ούτε